Οπότε θα γίνει έτσι σε αυτή την αλλαγή του ενός από την άλλη και τώρα επίσης προχωρούμε στην πρώτη ανάγνωση. Πρόκειται για τις θέσεις του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση και έχουμε επίσης τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει προθεσμία τριών μήνων. Στο τέλος του θα πρέπει από τις 24 Μαΐου και μετά θα αρχίσει να τρέχει η προθεσμία και μέχρι θα πρέπει να αποφασίσουμε και έχουμε το άρθρο 130 του κανονισμού σύμφωνα με το οποίο θέλω να σας προτείνω το πρώτο ε, μας σημείο εδώ που αφορά τις παραβίες των δικαιωμάτων να συζητηθούν όσον αφορά το τι έχει γίνει με τους κρατουμένους στο Γουεντάνομο. Αυτό θα πρέπει να ψηφιστεί χωρίς συζήτηση. Επίσης, σε ψήφιση θα θέσουμε την πρόταση αυτή. Θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τώρα